Good Γεια σας, <clears throat> κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Επόμενο θέμα στην εμεί διάταξη. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω τον κύριο Πέτερ Πελεγκρίνη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που είναι αρμόδιος για τις επενδύσεις και τη κοινωνία των πληροφοριών και ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας. Θα μας ενημερώσει και θα συζητήσουμε μαζί του αυτές τις προτεραιότητες. Όπως γνωρίζετε, στην αρχή κάθε Προεδρία του Συμβουλίου, ο αρμόδιος Επίτροπος για την Πολιτική Συνοχή έρχεται στην Επιτροπή μας για να εξηγήσει τις προτεραιότητες της νέας Προεδρίας του Συμβουλίου στους τομείς της δικής μας επαναλαμβάνω αρμοδιότητας. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Πελεγκρίνη και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, αναλαμβάνει σε πολύ δύσκολους καιρούς της ευρωπαϊκής ιστορίας και της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Σλοβακία. Εκτός από τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να αρχίζει να ασχολείται με τις συνέπειες των πρόσφατων αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προσπαθήσει να απαντήσει με τρόπο πιστικό στις επικρίσεις των λαϊκιστών. Αλλά εμείς έχουμε και την νομοθετική μας δουλειά που συνεχίζεται παρά αυτές τις προκλήσεις και τους χαλεπούς καιρούς. Και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω εξ όλων μας ευχόμενη πάρα πολύ καλή επιτυχία στη Νέα Προεδρία και πιστέψτε μας έχετε την πλήρη μας υποστήριξη. Προτείνω να ακολουθήσουμε τη συνήθη διαδικασία. Θα μιλήσει πρώτα ο Υπουργός, θα κάνει μια εισαγωγή και με περίπου 15 λεπτά, όχι παραπάνω, και μετά θα δίνω το λόγο στα μέλη για τις ερωτήσεις αρχής γενομένης από το γύρο των συντονιστών. Κύριε Πελεγκρίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της προτεραιότητες της Προεδρίας μας και το πρόγραμμά μας στην ε, πολιτική συνοχής. Η Σλοβακική Προεδρία, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, έρχεται μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και πρωτοφανή. Ε, η έκβαση του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο μας έχει φέρει ενώπιον νέων προκλήσεων. Για πρώτη φορά στην ιστορία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που ένα κράτος μέλος αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλαμβάνοντας λοιπόν την Προεδρία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν προβλήματα και κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει καλύτερη, ισχυρότερη και όσο γίνεται πιο ενωμένη όπου γίνεται αυτό. Εμείς θέλουμε να έχουμε θετικό πνεύμα και να λέμε πράγματα που καταλαβαίνουν οι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν κρίσιμο ρόλο εδώ να διαδραματίσουν στις δημοκρατίες μας και τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε εκλεγμένους εκπροσώπους 28 κρατών μελών ε, που τους έχει ανατεθεί ε, ε, αρμοδιότητα και δημοσιονομική αλλά και εποπτείας της νομοθεσίας. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο σας. Είχα την ευκαιρία και το προνόμιο να δω πολλά μέλη της Επιτροπής σας και θέλω να υπάρχει όσο γίνεται πιο αγαστή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και θα κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Επιτρέψτε μου τώρα να σας αναφέρω τις τέσσερις προτεραιότητες Σλοβακικής Προεδρίας. Μια Ευρώπη οικονομικά ισχυρή, σύγχρονη εσωτερική αγορά, ε, μια πολιτική ασύλου και μετανάστευσης βιώσιμη και μια Ευρώπη ε, παγκόσμια ε, πρωταγωνίστρια. Στην οικονομία τώρα, παρά τις κάποιες αναλαμβές ανάκαμψης, δεν έχει έρθει πλήρης ε, ανάκαμψη της οικονομίας. Πρώτη προτεραιότητα είναι να επικεντρωθούμε σε πρωτοβουλίες που ευνοούν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της Ένωσης. Η Προεδρία μας είναι πεπισμένη ότι η ε, χρηστή ε, χρήση των δημοσίων οικονομικών και οι μεταρρυθμίσεις οι διαρθρωτικές είναι στην καρδιά μιας ισχυρής Ευρώπης. Ο προπολογισμό του 2017 είναι άλλο σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό. Συχνά ε, αυτός ο κλήρος πέφτει στις προεδρίες του δευτέρου εξαμήνου. Η εσωτερική αγορά είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να ρίξουμε τους φραγμούς και να άρουμε τα εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια σφριγγυλή εσωτερική αγορά που θα είναι κινητήρας για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Θέλουμε να προωθήσουμε την Ενεργειακή Ένωση και την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά. Μετανάστευση. Ιστορικά είναι ένα φαινόμενο πανταχού παρόν. Οι σημερινέ μεταναστευτικέ ροέ όμω ε, πιέζουν περισσότερο τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν φιλοδοξία μας είναι η Ευρώπη να προχωρήσει προς μια πολιτική μετανάστευση και ασύλου βιώσιμη. Αφού λοιπόν τα έχουμε όλα αυτά στο εσωτερικό της Ένωσης, δεν μπορούμε να ξεχνάμε την συλλογική μας ευθύνη σε διεθνές επίπεδο. Η Προεδρία μας θα υποστηρίξει την ενίσχυση του παγκοσμίου ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τομείς όπως είναι η αναπτυξιακή συνεργασία, η Προεδρία μας θα επικεντρωθεί ε, στην εφαρμογή του θεματολογίου 2030. Μια που είμαι και στην Επιτροπή ε, για την Περιφερειακή Πολιτική, επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ. Η πολιτική συνοχής δεν ε, μειώνει μόνο τις διαφορές κάθε είδους, αλλά συμβάλλει και προς μια βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η πολιτική στο μέλλον υπό την Προεδρία μας θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής με νέα στοιχεία της μεταρρυθμίσης που θα τα αξιολογούμε και θα συζητήσουμε τις μελλοντικές προοπτικές. Έχει έρθει η ώρα να συλλέγουμε στοιχεία και να βάλουμε τα θεμέλια για τη μελλοντική συνεργασία. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη έχει ε, υποβληθεί μια πρόταση για τους μηχανισμούς από της Ελλάδας και της Κύπρου. Υπάρχει ευρεία στήριξη από τα κράτη-μέλη για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει σύντομα να καταλήξει σε κοινή θέση. Θέλουμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας για το θέμα αυτό και μάλιστα να το ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια της ε, Σλοβακικής Προεδρίας. Επιπλέον, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου ε, για ε, τα διαφθορτικά προγράμματα επετεύθη τέλος Απριλίου και τους επόμενους μήνες θα αρχίσουμε διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλη προτεραιότητά μας είναι η απλούστευση της πολιτικής συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση που έχει ε, εκδώσει μια σειρά συστάσεων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Μετά τις ελληνές διακοπές περιμένουμε νομοθετική πρόταση για την απλοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεργαστούμε στο Συμβούλιο αποτελεσματικά έτσι ώστε όλα αυτά το συντομότερο να εφαρμοστούν στην πράξη και οι διαχειριστικές αρχές και δικαιούχοι κοινοτικών κονδυλίων να δούνε πραγματικά ε, χειροπιαστά αποτελέσματα πολύ σύντομα. Βέβαια αυτέ οι αλλαγέ δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη σταθερότητα τη εφαρμογή ούτε να δημιουργούν, ε, να προκαλούν καθυστερήσει. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το μέλλον. Πώ ε, θα απλοποιήσουμε το εκτατικό σύστημα ελέγχου και να έχουμε περισσότερη προσέγγιση ε, στα αποτελέσματα. Θα χρειάζεται λιγότερο έλεγχο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Υπάρχουν ε, πολλές ευκαιρίες το για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Το Σεπτέμβριο 15 και 16 του μηνός θα έχουμε τη διάσκεψη για τη συνοχή στην Πρατισλάβα με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Κρέτσου και ελπίζω να παρεμβρίσκεστε και εσείς κυρία Μιχαήλοβα. Σε τρία πάνελ θα συζητήσουμε διάφορα στοιχεία ε, της πολιτικής συνοχής. Το πρώτο θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή των νέων στοιχείων της πολιτικής συνοχής το 2014-2020. Δεύτερο πάνελ. Σχέση ε, πολιτικής συνοχής και ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Και τρίτο πάνελ. Απλούστευση πέραν των τρέχουσών ε, προτάσεων και μελλοντικές διαδικασίες για την απλούστευση. Αυτό ήταν σημαντικό θέμα που κυριάρχησε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής περιφερειών και πόλεων στην Πρατισλάβα και όπου ήταν παρόντα και κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Επιτροπή των Περιφερειών και θα διοργανώσουμε ένα εργαστήρι για την απλούστευση και πάλι των χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης θα δώσουμε συνέχεια στο αστικό θεματολόγιο. Εγκρίθηκε στο Άμστερνταμ μια αστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς τώρα ερχόμαστε στην πρακτική εφαρμογή όλων αυτών. Η Σλοβακία μαζί με την πόλη της Βιέννης είναι ε, συντονιστής ε, για την εταιρική ε, σχέση για τη στέγη και τη στέγαση. Θα έχουμε και τρεις νέες συνεδριάσεις και υποστηρίζουμε τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που είναι τέσσερις. Έχουμε και τη στρατηγική του Δουνάβεως. Το πέμπτο ετήσιο φόρουμ θα το διοργανώσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 και 4 Νοεμβρίου και πάλι στην Πρατισλάβα. Αντίστοιχα με τις γενικές προτεραιότητες, το ετήσιο φόρουμ για το Δούναβι θα καλύψει θέματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, η κοινωνία της γνώσης, η διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ε, και ε, τα σχετικά. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 16 Νοεμβρίου που είναι αφιερωμένο στην πολιτική συνοχή, το Συμβούλιο Υπουργών θα ασχοληθεί με τα τρέχοντα νομοθετικά θέματα, την απλούστευση και την αξιολόγηση των νέων στοιχείων τη αναθεωρημένη πολιτική συνοχή. Εμεί θέλουμε να ακούσουμε με προσοχή, να φουγκραστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό το φθινόπωρο προγραμματίζουμε δύο εργαστήρια μαζί σα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με του Ευρωβουλευτέ. Το ένα για τι ευφύ πόλει και την ενεργειακή απόδοση και το δεύτερο για την εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία. Ελπίζουμε να είναι μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Really very much και προσβλέπω σε στενή και αγαστή συνεργασία μαζί σας και πιστεύω ότι αυτό ε, θα είναι ένα επιτυχές εξάμεινο προς όφελος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσουμε στους κοινούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Minister. Thank you for this presentation. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Θα ακούσουμε τώρα τους συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες. Βανίστερο από τα Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα θετική η προσέγγισή σας παίρνετε τη σκητάλη από τους Ολλανδούς και θα ολοκληρώσετε λέτε το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Ναι, να το ολοκληρώσετε, αλλά ε, ποια θα είναι η συμβολή σας για την πολιτική συνοχή. Θέλετε να αρχίσετε τους τριμερείς διαλόγους, όμως πρέπει να επιταχύνετε για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε σε σχέση με τα επιδιακόμενα αποτελέσματα. Είμαι λίγο σκεπτικός με αυτά που συνέβησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, κάποιες περιοχές πήραν τα περισσότερα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων δεν κατάφεραν ε, να μιλήσουν στις καρδιές ε, των ανθρώπων. Ενώ άλλοι ψήφισαν ε, θετικά όπως στη Σκοτία. Πρέπει να δείτε, να πάτε βαθύτερα, να έρθετε σε επαφή, να ε, εγκαθιδρύσετε μια σχέση με τους πολίτες. Είναι φούσκα εδώ. Εμείς είμαστε μέσα σε αυτή τη φούσκα των Βρυξελών. Η δουλειά μας είναι όμως να έχουμε μία ισορροπία στην Ευρώπη. Κυρίως για θέματα εδαφικής συνοχής. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, τι θέλετε να επιτύχετε ακριβώς, πιο συγκεκριμένα μπορείτε να μας το πείτε, σε σχέση με την πολιτική συνοχή γιατί δεν το ακούμπησαν οι Ολλανδοί. Μία διάσκεψη έκανα σε επίπεδο διευθυντών και δεν εδόθη συνέχεια. Η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία από οικονομικής πλευράς ήταν το βασικό. Το μέλλον της συνοχής δεν το άγγιξαν καθόλου. Είστε ιδανικοί για να το κάνετε και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από σας οι χώρες ε, Βίζεγκρατ κατέθεσαν ήδη τις ιδέες τους και όταν τις διαβάζω βλέπω μία εγκύτητα σε σχέση με τις φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές προοπτικές. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος λοιπόν. Μετά ζητάτε ανοιχτό διάλογο πολύ καλά και χαιρόμαστε που θα έρθετε για διάφορα εργαστήρια και σεμινάρια. Και αυτή Μήπως θα έπρεπε να ε, μας στείλετε περισσότερες προσκλήσεις για την διάσκεψη το Σεπτέμβρη, για να έρθουν όσο δυνατόν περισσότεροι βουλευτές, γίνεται. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα να πω. Α, ναι, και για το μέλλον... Καλό θα ήταν να μην μιλάμε μόνο για κατανομή κινδύνου και ευθυνών. Τώρα με το έτσε έχουμε ε, έχουμε ουρεάνεμο. Όμως μετά θα πείτε, πρέπει να αποπληρωθούν τα δάνεια. Δίνουμε τόσα ε, ε, σε αυτό το πρόγραμμα και μετά από μία δεκαετία περιμένετε να πάρετε πίσω τα λεφτά. Για τους μετανάστες, για πρόσφυγες, για τέτοια. Δεν γίνεται να το ζητάτε αυτό. Χρειάζεται επιδοτήσεις. Γιατί στο FC ωραία το έχουν βρει, έχουν αλακάρτε διαλέξει ό,τι θέλουν από τα προγράμματα, αλλά δεν έχουν όμως ε, ολιστική προσέγγιση. Εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε οι πόλεις, οι περιοχές με ολιστικό τρόπο να συνεργαστούν, ούτως ώστε να μπορέσουμε εμείς να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Εσείς πώς τοποθετήσετε. Ευχαριστώ και πάλι από πλευρά του που ήρθατε. Σοσιαλιστές, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πελεγκρίνη για τις παρουσιάσεις σας αυτές. Πρέπει να πω ότι αν δεν υπήρχε το βρετανικό δημοψήφισμα, είναι καταπληκτικό το πρόγραμμά σας. Δεν φταίτε εσείς τώρα βέβαια που 7 μέρες πριν αρχίσει η προεδρία σας έχει το δημοψήφισμα αυτό με το γνωστό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε εμείς ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στο Συμβούλιο να συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Και μάλιστα τώρα ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις που κάποια στιγμή θα αρχίσουν αναγκαστικά και ανεξάρτητα τελείως επίσης από όλα αυτά θα πρέπει να είναι φιλοδοξία και αξίωση της δικής σας Προεδρίας να κοιτάξετε πώς μπορούμε να ανακτήσουμε ε, λίγη από αξιοπιστία και εμπιστοσύνη που δεν έχει να κάνει μόνο με το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό, είναι και πανευρωπαϊκό. Και πραγματικά θα επιθυμούσα, τουλάχιστον παράλληλα με τη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, να γίνει και μια άλλη. Για το πώς, για παράδειγμα, ε, προβάλλουμε την πολιτική συνοχή στα κράτη-μέλη. Καμιά φορά συμβαίνουν εδώ πιστήρια πράγματα μας ζήτησε ένα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη-μέλη να διαφημίζουμε περισσότερο το σχέδιο Juncker στις περιφέρειες για να πετύχει. Ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά. Και καλά τα λέει ο Αντιπρόεδρος, αλλά θα το κάνουμε προφανώς ως βουλευτές. Αλλά δεν μπορούμε να βγαίνουμε μόνοι μας και πλασιέ σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε διαφήμιση ότι κοιτάξτε υπάρχουν τα διαρθρωτικά ταμεία, ότι πετύχαμε πάρα πολλά σε, πολλά, σε όλα τα κράτη-μέλη. Επιτέλους θα πρέπει να το λένε και τα ίδια τα κράτη αυτά και να τα διαφημίσουν. Και εγώ θα επιθυμούσα η Σλοβακική Προεδρία να το συμπεριλάβει ως ένα επιπλέον στόχο. Γίνεται αυτό, να προσθέσετε και άλλο στόχο. Αν καταφέρουμε να τα επικοινωνούμε αυτά διαφορετικά στα κράτη-μέλη, τότε θα ήταν ήδη τεράστια επιτυχία. Συμφωνώ μαζί σας ότι χρειαζόμαστε μια συγχρονή εσωτερική αγορά για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αλλά τι να την κάνω την εσωτερική αγορά αν δεν θέλει κανένας να συμμετέχει. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό πραγματικότητα να σηκωθεί να φύγει γιατί το θέλει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα όμως που συνέβη το μοιραίο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ακολουθήσουν και άλλα κράτη. Και πώς θα γίνει αυτό. Αυτό γίνεται όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου αλλά και όταν το λες για να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Θα μπορούσατε να του συμπεριλάβετε και αυτό στο σχεδιασμό σα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Μια πολύ σύντομη ερώτηση οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, ε, σύγχρονη ενιαία αγορά, καλή πολιτική ασύλου, ε, η Ευρώπη ως παγκόσμιος επέκτης ε, και η πολιτική συνοχή είναι η κόλλα που τα κρατάει όλα αυτά ενωμένα. Μπορείτε να πείτε λίγα περισσότερα για την σύγχρονη ενιαία αγορά. Ευχαριστώ, μου από τη Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε ως μέλος του Ολλανδικού Κοινοβουλίου είμαι... Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαι πεπισμένος ότι θα ε, καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχει επιτυχία η Προεδρία σας. Κάνατε πολλά για το αστικό θεματολόγιο και από ό,τι κατάλαβα θα συνεργαστείτε για αυτό συγκεκριμένο φάκελο με την Ολλανδική Κυβέρνηση. να συγχαρώ για τη δουλειά που κάνετε στο τρίο της Προεδρίας και είναι πολύ καλή ε, αυτή η χειρονομία πλευράς Ολλανδικής ε, κυβέρνησης να συνεργαστεί μαζί σας. Μπορείτε να επεκταθείτε γιατί το πρόγραμμα σας, μιλήσατε για τη γέννα, για τη στέγη, στέγα, τα προγράμματα στεγαστικά και με την Προεδρία της Μάλτας και την επόμενη θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα ε, της ανάπτυξης των αστικών περιοχών. Το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον είναι η μετανάστευση. Η συνοχή σημαίνει και αλληλεγγύη και ε, αφήνουμε τις μεγαλόσχημες δηλώσεις, αφήνει το Συμβούλιο τις μεγαλόσχημες δηλώσεις ε, και βάζει λεφτά, κυρίως ε, εκεί που χρειάζεται για τους πρόσφυγες τα μέσα τα δίνει η πολιτική συνοχή για να γίνουν επενδύσει για την ε, ενσωμάτωση των προσφύγων σε πολλές χώρες. Θα τηρήσετε τα υπεσχημένα στο Συμβούλιο, πρώτη ερώτηση, για το κονδύλι για τους πρόσφυγες και θα έχει το σωστό μείγμα των ε, μέσων της πολιτικής συνοχής για να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τους, ώστε και στη Σλοβακία να σωματωθούν στην κοινωνία οι πρόσφυγες και να δώσετε το παράδειγμα ίσως στην Ευρώπη. Ε, σας ευχαριστώ και τον προτείνω για τις απαντήσεις σας και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Βάνα Πράσινη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε και σας ευχαριστώ για την προσφορά σας για στενή συνεργασία το επόμενο εξάμεινο. Θέλω να πω κάτι θετικό. Έχετε πιο ειδικό πρόγραμμα για την πολιτική συνοχή από ότι ε, στο πρόγραμμα το γενικό της Σλοβακικής Προεδρίας. Στη σελίδα 13 είδα μόλις μια μικρή αναφορά γενικά για την πολιτική συνοχή. Και εδώ είπαν και οι προλαλήσαντες ότι το επόμενο εξάμεινο πρέπει να μπει πιο ψηλά στις προτεραιότητες η πολιτική συνοχής λόγω και των προσφάτων εξελίξεων. Πάντως σας πιστεύω ότι προσωρινά, μάλλον προσωπικά θέλετε να δώσετε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, είπε και ο προλαλής κάτι. Θέλω να ρωτήσω για τους πρόσφυγες, δεν θα το επαναλάβω, τα ίδια με τον προλαλήσαντα. Η ε, πολιτική για τους πρόσφυγες είναι μία από τις προτεραιότητες, έτσι δεν είναι. Και εμείς αγωνιστήκαμε πολύ τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία να ανοίξουν ακριβώς για μέτρα υπέρ της ένταξης των προσφύγων, ιδιαίτερα το Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΤΠΑ, το Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αλλά γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν το δέχονται πάρα πολύ προώθημα αυτό. Η δική σας Προεδρία του Συμβουλίου δεν θα μπορούσε κάπως να παροτρύνει τα κράτη-μέλη. Όπως είπε και η κυρία Κρέλ, εμείς ως απλοί ευρωβουλευτές δεν μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή την επικοινωνία και την προβολή ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες. Πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, όσα τους αναλογούν. Και ιδιαίτερα στο προσφυγικό θα πρέπει να ε, εμφανιστούν όχι απλώς για την κατανομή των προσφύγων αλλά και γενικότερα για να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που υπάρχουν. Ακούμε συνέχεια δεν έχουμε λεφτά. τώρα έχουμε γιατί δεν τα δαπανούν τα κράτη-μέλη. θα αναλάβετε τέτοια πρωτοβουλία. Δεύτερη ερώτηση. Πολύ θετικά επίσης σημείωσα αυτά που είπατε για την Urban Agenda, το αστικό θεματολόγιο, πολύ ωραία, και για τη δική μας επιτροπή γυριάρχησε αυτό το θέμα, ήταν και έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας αυτή που εγκρίναμε για να αναγνωρίζονται περισσότερο οι πόλεις. Εγώ ξέρετε είμαι Βιενέζα και ε, στα θέματα της στέγης ε, Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια, αλλά είναι τέσσερις οι προτεραιότητες για το θεματολόγιο αυτό, το αστικό, είναι ο ατμοσφαιρικός ε, αέρας, η φτώχεια, η μετανάστευση και η στέγαση. Αυτά είναι τα τέσσερα. Το ίδιο πρόβλημα το έχουμε ε, και με τα κράτη-μέλη. Τα προγράμματα των πόλεων για καινοτόμες δράσεις, ε, για τους πρόσφυγες, την χάνουν χείρις της από τον τόπιο πληθυσμό. Αυτό είναι δική σας προτεραιότητα. Thank you very much. I have three more names. Ευχαριστούμε. Άλλοι τρεις είναι στον κατάλογο για τις ερωτήσεις. Τέσσερις τώρα. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό, όμως πρώτα για κάποιες απαντήσεις και μετά συνεχίζουμε, κάνουμε δεύτερο γύρο. Ωραία. Θα μιλήσω τη μητρική μου, αν δεν σας πειράζει, ε, για τις απαντήσεις. Ελπίζω να με μεταφράσουν. Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας. Κάποιες μπορώ να τις ομαδοποιήσω. Κάποιες θα τις απαντήσω μεμονωμένα σίγουρα. Κύριε Βανίστεροι και κυρία Κρέλ. Είναι δύσκολο να ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της δουλειάς μας όχι μόνο σε σχέση με το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχουμε την εντύπωση πως Οι πολίτες δεν συνειδητοποιούν τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη χώρα τους. Αποφάσισε μια χώρα να αποχωρήσει. Αυτό νομίζω θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για να επανασχεδιάσουμε την προσέγγιση μας και να έχουμε ενότητα. Σίγουρα δεν θέλουμε τώρα να ε, αρχίσει ένα κύμα αντίστοιχων αντιδράσεων σε άλλες χώρες. Γι' αυτό, μιλώντας για την πολιτική συνοχής, στη Σλοβακία τουλάχιστον ε, δεν είναι ευνόητη η πολιτική συνοχή για τον πολίτη. Πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα των πολιτών. Να γίνουμε κατανοητοί. Δηλαδή, να βασιστούμε σε συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα αποτελέσματα ανά χώρα, πώς βελτιώσαμε την υποδομή, πώς βελτιώσαμε τη στέγαση και ούτω καθεξής, να τα παρουσιάσουμε ως αποτέλεσμα της αλληλεγγύης που δείχνουν τα πιο προηγμένα κράτη προς τα λιγότερο προηγμένα. και να ξεκαθαρίσουμε ότι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε δυνατή την ε, εφαρμογή, την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Ούτε πρέπει να θεωρούν δεδομένο το μέλλον οι πολίτες θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο που χαράξαμε. Σίγουρα θυμούνται κάποιοι τα σύνορα που είχαμε στην Ευρώπη. Κάποιοι θεωρούν δεδομένη ελεύθερη κινητικότητα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε καν μπορούν να διανοηθούν πώς θα ήταν να ζουν χωρίς το Σέγγεν. Ανοιχτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε την ε, επίγνωση των πολιτών ε, για τα πλεονεκτήματα μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συνοχής έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, όμως είναι εξαιρετικά κακή η φήμη της. Πάντοτε αναφέρεται η πολιτική συνοχή ε, σε αρνητικά συμφραζόμενα. Όλοι και στα κράτη-μέλη και οι βουλευτές του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διαδίδουν τα ωφέλη και τα καλά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Βρίσκω πως είναι ιδιαίτερα επικοδομητική η προσέγγισή σας. Διότι έχετε ένα όραμα για το μέλλον πέρα από το δημοσιονομικό κομμάτι του τομέα. Κύριε Φανιστερόε, ε, με ρωτήσατε τι θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Έχει υπογραφεί η συμφωνία, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, όμως ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται στο σύμφωνο. Αυτό το αστικό θεματολόγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το τέλος της διαδικασίας, είναι απαρχή μιας διανέας διαδικασίας. Πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το δρόμο που χαράξατε. Δεν θέλουμε να οργανώσουμε μόνο συζητήσεις, διασκέψεις και να κινούμαστε σε θεωρητικά επίπεδα. Θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν διαπιστώνουμε ότι χωλαίνει ένα πρόγραμμα, δεν είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να διαπιστώσουμε σε τι οφείλεται αυτό για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Για την απλούστευση, πέρα από την ε, περίοδο μέχρι το 2020, θα πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα προγράμματα ανά κράτος, να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ότι είμαστε μεταβατική περίοδο ανάμεσα σε δύο ε, διαδοχικές ε, προγραμματικές περίοδους. Και ως εκ τούτου έχουμε και αυξημένο γραφειοκρατικό φορτίο είναι και αυτό μια πρόκληση. Θα τέλη του 16 και στις αρχές του 17 θα καταφέρουμε να ε, αυξήσουμε τις επιδόσεις των προγραμμάτων. Σίγουρα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για την απλούστευση. Αυτό επιδιώκουμε. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε πολυσέλιδα ογκώδη έγγραφα που θα περιπλέξουν την περαιτέρω τη διαδικασία. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Θέλουμε αυτά αποτελέσματα και που δεν είναι άρδινα αναθεώρηση του τρόπου εργασίας. Θέλουμε άμεσα αυτά αποτελέσματα. Ε, θα ήθελα να περάσω τώρα στην άλλο σημείο. Πανάκτηση της εμπιστοσύνης και σε αυτό το τομέα. Έχω την εντύπωση ότι δεν συνεργαζόμαστε όλοι πάντοτε ικανοποιητικά εννοώ τα, ε, όλα τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και οι πολίτες, θα πρέπει να κοιτάζοντας τις περιοχές να βλέπουμε υπόπτους, ε, να φοβούμαστε ότι θα κατασπαταλήσουν το δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να ε, τους έχουμε εμπιστοσύνη, να έχουμε εμπιστοσύνη στην υπεύθυνη προσέγγιση που θα υιοθετήσουν Ε, για την χρήση αυτών των κονδυλίων, όπως τους έχουμε εμπιστοσύνη και για τους φόρους που συλλέγουν. Όταν υπάρχουν πάντοτε υπόνοιες και υποψίες για διασπάθηση, τότε ε, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Ε, και μεταξύ άλλων, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνη έχουμε ε, μια ένα ολόκληρο πλωστάσιο περίπλοκους κανόνες. Λοιπόν, θα πρέπει να απλωστεύσουμε τις διαδικασίες, δώσω την η πολιτική συνοχή, του μέλλοντος να είναι απλούστερη. Αυτό μπορούμε να συζητήσουμε μετά το 2020. Πώς γίνεται, πώς θα μπορέσει να αναβαθμιστεί αυτή η πολιτική συνοχή. Δεν χρειαζόμαστε ριζοσπαστικές αλλαγές. ούτε αλλαγή πορείας. Περισσότερη διαφάνεια χρειαζόμαστε και να καταλάβουμε πώς θα συνδυάσουμε αυτή την προσέγγιση με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Κύριε Βανίστερο, συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλες τις επιδοτήσεις. Τις δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούμε όλες να τις χρηματοδοτούμε με αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Συμφωνώ. Για τη διαχείριση του χρέους ε, οφείλουμε να υπακούσουμε σε διάφορους κανόνες και ξαναλέω θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορες μορφές στήριξης. Κύριε Τόμας έτσι. Εσείς ρωτήσατε για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα έχω λοιπόν την τιμή αύριο σε μια άλλη επιτροπή να σας παρουσιάσω ολόκληρο το πρόγραμμά μας σε αυτό το θέμα. Θέλω εντάχει να σας πω περί τίνος πρόκειται, η ψηφιακή αγορά είναι προτεραιότητα για μας. Μετά την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών υπηρεσιών και προσώπων, θεωρούμε πως η ελεύθερη μεταφορά, μετακίνηση δεδομένων είναι βασική ελευθερία. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει ομοιομορφία ως προς την κανονιστική ρύθμιση. Έχουμε 28 Μονομένε αγορές και σύνορα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, σκοπεύει να γίνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας. Θα θέλετε λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα, με τα χαράς να σας τις δώσω αύριο στην παρουσίαση. Κύριε Βίλτεμπουργκ, ζητώ συγγνώμη, δεν εκπροσωπώ την Σλοβακική Δημοκρατία εδώ σήμερα. Δεν υπεραμείνω με τις ε, θέσεις της χώρας μου για το μεταναστευτικό εκπροσωπώ το Συμβούλιο για την ε, πολιτική συνοχή σε αυτή τη στιγμή, κύριε Βαν Μίλτεμπορκ. Ο καθένας ε, μπορεί να αποκομίσει διαφορετικές ε, εντυπώσεις σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολύ θετικές δράσεις σε συνεργασία με την Αυστρία. Δεν θα ε, σχολιάσω άλλο αυτό το ζήτημα γιατί δεν είναι της παρούσης. Κύριε Βανά, μιλήσατε για τη χρήση των κονδυλίων, ε, για το, το μεταναστευτικό, για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων. Σίγουρα ε, θέλουμε, αν τα κράτη-μέλη το επιθυμούν, να χρησιμοποιήσουμε μονομενα επιχειρησιακά προγράμματα, ούτως ώστε να θέσουμε στη διάθεσή τους κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιήσουν ε, κατά ε, ε, το δοκούν. Έτσι, μπορεί να, μπορούμε να μεταφέρουμε τα κονδύλια σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο αποτελεσματική έτσι, η διαχείριση των κονδυλίων που θα έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επαρκή πρικοδότηση από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και από τα υπόλοιπα ε, χρηματοδοτικά μέσα για να μπορέσει να ε, έχει την κατάλληλη απόκριση στις κρίσεις. Δεν μπορούμε από την πολιτική συνοχή να βρίσκουμε τα επιπρόσθετα κονδύλια. Θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τον προπολογισμό. Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν εδώ και 10 χρόνια. Τότε ήταν προτεραιότητα. Όχι πλέον απαραίτητα σήμερα όμως. Τους πόρους να τους ψάξουμε λοιπόν σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού. Και όχι να παίρνουμε χρήματα μόνο από την πολιτική συνοχή κάθε φορά που ε, προκύπτει μια κρίση. Για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων ε, έχουμε στην αγορά εργασίας διάφορα εργαλεία για την ε, ε, καλύτερη κατάρτιση για την ε, απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Όλα αυτά μπορεί να τα καλύψει το ΕΚΤΕ. Η Σλοβακία αυτό το δρόμο ακολουθεί ήδη. Σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε διεξοδικότερα αυτό το ζήτημα και συντρέχουν όλες οι προποθέσει για να γίνει πολύ υπεύθυνη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Κύριε Πελεγκρίνη, σα ευχαριστούμε. Θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Μικουλάσιτς θα πάρει το λόγο. Το είπα καλά. You said very correct. Ναι, πολύ σωστά. Ε, κάποιοι με φωνάζαν και Μιλόσεβιτς παλιότερα, αλλά δεν είναι το όνομά μου αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Ρέτζι στο Ευρωκοινοβούλιο ε, και εγώ χρησιμοποιώ την γλυκιά μου μετρική γλώσσα για να... και θα με καταλάβετε έτσι καλύτερα νομίζω. Οι παρατηρήσεις μου στόχο έχουν να είναι επικοδομητικές. Ο συνάδελφος Βανέστε Ρόι, αλλά και πάνω απ' όλα οι φίλοι η Κωνσταντζα Κρέλα, Μίλησαν για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Ε, Επίση, ε, στην Ευρώπη υπάρχουν ε, πολλοί νέοι που δεν ξέρουν πια ε, ούτε πού βρίσκονταν τα σύνορα. Η Σλοβακία δυστυχώς ε, είναι διάσημη διότι στις τελευταίες δύο εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο είχε τη μικρότερη συμμετοχή ε, στις ευρωεκλογές. Είναι λυπηρό, είναι απίστευτο. Κάτω από το 20% συμμετοχή σε τελευταίες ευρωεκλογές δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Και γιατί είναι έτσι, γιατί είναι, είναι το μέλλον. κάτι στο οποίο θα έπρεπε να στοχεύουμε. Ε, το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολύ επιφανειακές πληροφορίες και ε, κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πάντα. Θα έχετε ακούσει και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό Φίτσο στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα να κάνουμε έναν παραλληλισμό, αν μου επιτρέπετε. Ο David Κάμερον για έξι χρόνια ήταν ε, πρωθυπουργό και επέκρινε τις Βρυξέλλες. Ε, οι Βρυξέλλες είναι ε, κακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας, τους Βρετανούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσάρεστη κτλ. κτλ. Και μετά, τρεις μήνες πριν από το Brexit, ξαφνικά άρχισε να λέει τι καλή που είναι η Ένωση και να γίνεται το συνήγορο του Remain και να μείνουμε στην Ένωση. Κανείς δεν κατάλαβε τι γινόταν βέβαια γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγε το τελείως αντίθετο. Εσείς είστε πολύ ικανός άνθρωπος και θέλω να σας ζητήσω το εξής και μέσω ημών και τον ε, Σλοβάκο Πρωθυπουργό. Έχουμε κατασκευάσει αυτοκινητοδρόμους, ε, αλλά λέτε και περαφανεύεστε γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν λέτε ότι αυτά έχουν γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα. Λέτε ζήτω, φτιάξαμε αυτό, αλλά ποτέ δεν λέτε ότι συμμετείχαν οι κονδύλια συνοχή. Αν μπορούσατε να το κάνετε αυτό κάθε φορά και να λέτε και να ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμο αλλιώ αντιλαμβανόταν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι είχα δίκιο, γιατί έκανε αυτή την παρατήρηση και στην Ολομέλεια την περασμένη φορά. Και ο Πρωθυπουργό σα είπε λοιπόν ότι είχα δίκιο και άρχισε να απαντά άλλο, σε άλλο τόνο. Το 86% των επενδύσεων που γίνονται στη Σλοβακία, αν σκεφτούμε αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους κτλ, το 86% λέω είναι από τα ευρωπαϊκά χρήματα. Εγώ ίδιος ε, ε, έχω ζήσει στο Κίσουτς, μια πολύ πολύ φτωχή περιφέρεια. Και τι έγινε σε αυτή την περιοχή, έξι μεγάλα project ε, που κατασκευάστηκαν χάρη στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η, προσέλευση στις ευρωεκλογέ ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Άρα το μήνυμα δεν περνάει. Και θέλω να σας καλέσω και σας προσωπικά, κύριε ε, Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, και να καλέσω γενικά τη Σλοβακική Προεδρία να βρει τη σωστή γλώσσα, ώστε το μήνυμα να φτάνει και στον ε, κάθε πολίτη, στον κάθε ψηφοφόρο. Για να καταφέρετε αυτόν τον απλό στόχο, τι κάνετε λοιπόν. Κάτι ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ε, ξεχάσατε κάτι. Δεν ξέρω αν οφείλεται αυτό στα όσα είπε η κυρία Κρέτσου ή στις παρτερίσεις, ε, κάποιων χωρών. Εν πάση περιπτώσει, στρατηγική για τα Καρπάθια. Ε, υπάρχει μια στρατηγική για την Καρπάθια, μια για το, ε, το Ιόνι, μια για την Αδριατική, μια για το Δούναβι, μια για τη Βαλτική. Θα... Εντάξει, σίγουρα και η Σλοβακία και άλλες περιφέρειες μπορούν να ωφεληθούν από τη στρατηγική για το Δούναβι, αλλά προς τα ανατολικά είναι οι πιο φτωχές περιφέρειες, οι πιο φτωχές περιοχές. Το ΑΕΠ κατά κεφαλή είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το μέσο όρο της Ένωσης. Ε, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ανατολική Τσεχία, η Σλοβακία και όλες αυτές οι χώρες. Λοιπόν, αυτή η στρατηγική για τα Καρπάθια που αφορά όλες αυτές τις χώρες δεν φαίνεται να απασχολεί κανέναν άλλον εκτός από την Πολωνία. Κανένας δεν ασχολείται με το θέμα της στόχιας. Εγώ πιστεύω πως οι ε, πολίτες θα πρέπει να βοηθηθούν και δεν μιλώ για νέα χρήματα, νέα κονδύλια. Φτάνει να ανακατανεμηθούν αποτελεσματικά μέσω μιας μόχλευσης, για παράδειγμα, τα χρήματα που υπάρχουν. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να προσεχθεί. Ευχαριστώ. Κυρία Σμάλκοβα, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Περεγκρίνη, δεν κρύβω ότι γνωριζόμαστε πάνω από 17 χρόνια. Ήμασταν ε, βουλευτές ε, καθομαστε διπλα δίπλα-δίπλα στο Κοινοβούλιο της Σλοβακίας γνωρίζω την υπευθυνότητά σου και την αποφασιστικότητά σου και είμαι βέβαια ότι τα όσα μας ε, παρουσίασες ως πρόγραμμα θα υλοποιηθούν και θα το τσεκάρουμε το Δεκέμβριο και είμαι βέβαια και ότι θα δοθεί όθηση στην πολιτική συνοχή. Εγώ έχω να κάνω μια παρατήρηση που προέρχεται από το γεγονό ότι χωρίς ε, τη διευθυντικά ταμεία η δική μου περιοχή, η Ανατολική Σλοβακία δεν θα είχε ούτε ένα βήμα μπροστά. Έχουμε ένα σωρό μικρά χωριουδάκια 100-200 κατοίκων όπου ο δήμαρχος ε, δουλεύει ε, κατά το 1 τρίτο στη δημαρχία. Και τα διευθυντικά ταμεία λοιπόν χρησιμοποιούνται αξιοποιούνται. Όμως χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά από πλευράς αυτών των μικρών ε, μονάδων. Ίσως ο κάποιος να ξέρει να κάνει κάτι, αλλά αν ο δήμαρχος δεν καταλάβει κάτι, μπορεί να χαθούν τελείως τα κονδύλια. Αυτός, η, αυτός ο, αυτή η πολιτική συνοχή μας επιτρέπει σιγά σιγά να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μπορέσουν να ζητήσουν χρήματα όλοι αυτοί οι μικροί δήμοι. Γιατί αν κάποιος κάνει ένα αίτημα ε, και απορριφθεί το αίτημά του, μετά μπορεί να μην ξανακάνει. Εγώ το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, διότι η διαδικασία είναι πολύ βασανιστική. a možno aj na eh, eh, Χρειάζεται λοιπόν να απλοποιηθούν τα πράγματα, κυρίω για τι πιο απομονωμένες περιοχέ, γιατί συχνά υπάρχουν ομάδε ε, όπω οι ευρωσκεπτικιστέ. έχουμε και έναν εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο από τη Σλοβακία, και που θέλουν να απομακρύνουν ακόμα περισσότερο αυτές τις ε, απομονωμένες ορεινές περιοχές, να μην δώσουν Ε, τίποτα, αλλά εμεί δεν θέλουμε να δώσουμε αυτό το είδο ε, τη λαβή. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωή στι ορεινέ και απομακρυσμένε περιοχέ, πρέπει και να τι βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την περιφερειακή πολιτική και αυτό την έκκληση κάνω προς την ε, Προεδρία ώστε να γίνουν σταδιακά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ωραία η τοποθέτησή σας κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης το πρόγραμμά σας, για να με δεν το διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι το θέμα της ε, περιφερειακής πολιτικής το έχετε δει λίγο ξόφαλτσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας σας. Άκουσα αυτά που είπατε ξεκαθάρισε ε, στο μυαλό μου αυτό που εννοεί η Σλοβακική Προεδρία. Ωραία. Θα ήθελα να κάνω ερωτήσεις για δύο τομείς. Και συνεχίζω από εκεί που ε, σταμάτησε η προλαλή σας. Τι γίνεται με τον κοινό σχεδιασμό. Αυτό το εργαλείο δεν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Καμιά φορά το λησμονούμε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά παραδείγματα για συνεργασία και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να υποστηρίξει ε, την ανάπτυξή του με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να χρησιμοποιείται αυτός ο μηχανισμός πιο συχνά. Πράγμα που σήμερα δεν συμβαίνει. Ακούγοντας λοιπόν όλους τους συναδέλφους, τι διαπιστώνω, ότι η Ευρώπη είναι πολύ άγνωστη. Ε, τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν φτάνουν στους πολίτες, δεν το συνειδητοποιούν οι πολίτες, δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα ωφέλη προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι λέμε συχνά. Ότι ε, η επιτυχία έχει πολλούς ε, πατέρες, ενώ η αποτυχία είναι ορφανή. Θα πρέπει λοιπόν η επιτυχία να προβάλλεται για να το μαθαίνουν οι πολίτες. Ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και της επιλογής των έργων που υποστηρίζονται. για να πιάνουν τόπο τα κονδύλια και να το ξέρουν όλοι. Να ξέρει ο καθένας πού πηγαίνουν τα κονδύλια. Και οι πολίτε. Για να μην βγαίνουν και λένε εκ των υστέρων οι πολίτες ότι δεν ξέραμε τίποτα και τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. σε όλα τα προγράμματα, σε όλα τα έργα να ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα ποιος πληρώνει τι και ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Πολύ συγκεκριμένες σκέψεις είναι αυτές. Και ε, σε σχέση με το Βρετανικό δημοψήφισμα. Βλέπουμε ότι οι περιφέρειες στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν ευεργετηθεί, ε, που έχουν ρεύσει τόσα κονδύλια, ε, ψήφισαν υπέρ του Brexit, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πολλά από τα έργα αυτά είναι άγνωστα. Είναι τεράστια η αποξένωση και η απόσταση που μας χωρίζει από τους πολίτες. Και μάλιστα όχι ότι υπάρχει ένα έργο που το χρηματοδοτεί η Ένωση, να ξέρουμε και τι κάνει. Μάλιστα, θα ήθελα και ο κύριος Φανίστερο να πει δύο λόγια, μόνο δύο. Ρώτησα κάτι για τη συμμετοχή μας. Εδώ βλέπουμε στο κατάλογο 15 και 16 Σεπτεμβρίου, το είπατε και εσείς, και μετά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Για τα αποτελέσματα και τι θέλετε να πετύχετε. Ε, εδώ μιλάμε για το μέλλον της συνοχής και είναι η ώρα των αποτελεσμάτων αυτή και των συμπερασμάτων τον Νοέμβριο. Και θα μας καλέσετε και μας εκεί και μπορούμε να συμμετέχουμε. Υπάρχει ευκαιρία για συζήτηση και με εμά δηλαδή ή γενικώ μεταξύ σας θα τα λέτε. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Thank you. These were more than two. Μόνο δύο λόγια δεν ήταν, αυτά ήταν παραπάνω. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά ήθελα να πω. Ωραία, μπορείτε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσω με τη σειρά. Κύριε Μικολάσεκ, σας διαβεβαιώ ότι προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να βελτιώσουμε την ε, εγρήγορση των πολιτών και την ε, συνειδητοποίηση. Έχουμε αυτή τη θλιβερή πρωτιά στη μεγαλύτερη αποχή στις ευρωεκλογέ στη Σλοβακία. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι τα ε, πράγματα παρουσιάζονται διαφορετικά από αυτά που είπατε και στον τύπο και ο Πρωθυπουργό μα μίλησε για σημαντικά έργα και για τον σημαντικό ρόλο τη πολιτική συνοχή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι έτσι όπω τα λέτε. Εμεί καταθέσαμε τις προτάσεις, παρουσιάσαμε την πολιτική συνοχή όταν εγκαινιάσαμε τη νέα γραμμή του τραμ στην Πρατισλάβα. Ή εχθές που δόθηκε στην κυκλοφορία ένα τμήμα αυτοκινητοδρόμου με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αλλάξει η γλώσσα που χρησιμοποιούμε λοιπόν και στη Σλοβακία και τα προβάλλουμε αυτά βεβαίως και τα διαφημίζουμε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ε, απλώς θέλω να πω ότι τα θέματα που μας απασχολούν ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είναι και νομοθετικού και μη νομοθετικού χαρακτήρα. Θα πρέπει τώρα να καταβάλουμε ε, και νέες προσπάθειες για να συμπεριλάβουμε τα νέα δεδομένα στη δουλειά μας. Να επιστρέψουμε στα βασικά, στα θεμελιώδη, back to basics, να χρησιμοποιούμε μια ε, γλώσσα πιο εύληπτη από τους πολίτες και από τους νέους. Να είναι πιο sexy, και το λέω έτσι ίσως προκλητικά, αλλά να είναι πιο ελκυστική η γλώσσα μας. Το είπε και ο κύριος Πότσακ. αν θέλεις να ενημερώσεις τους πολίτες για ένα έργο και για ένα πρόγραμμα, δεν αρκούν τα πανό και ε, οι αφήσει με τα στεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζονται νέες τεχνολογίες, σύγχρονες, τα social media. Από εκεί επικοινωνούν οι νέοι. Αυτές είναι οι πλατφόρμες. Εκεί βρίσκεται ο κόσμος ο νέος. Και θα πρέπει να συζητάμε και να προβάλλουμε αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Γιατί καμιά φορά είναι γεγονός αυτό σε εθνικό επίπεδο. Οι Βρυξέλλες είναι βρισιά. ανάλογως με τα συμφέροντα κάποιου πολιτικού ε, κόμματος. Ε, μιλήσατε για ένα μικρό χωριό. Ναι, το είπαμε και στη Σύνοδο Κορυφής των Πόλεων και των Περιφερειών. Υπάρχουν ε, μικρές δομές, μικρές ε, πόλεις ή μικρά έργα που δεν ε, ζητούν χρηματοδότηση, δεν καταφεύγουν σε αυτή τη δυνατότητα γιατί είναι τεράστια επιβάρηση γραφειοκρατική και άμα ζητήσουν και λογιστικό έλεγχο από δύο λογιστές μπορεί να καταλήξουν και σε διαφορετικά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν η λογοδοσία να υπάρχει αλλά να γίνεται με πιο απλό τρόπο, με συγκεκριμένες μεθόδους. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα χρήματα αυτά έρχονται από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Δεν είναι δικά μας, ούτε δικά σας. Είναι των Ευρωπαίων φορολογουμένων που οι περισσότεροι ζουν σε ευρωπαϊκές πόλεις και χωριά. Άρα θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε και τα ωφέλη για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα πρέπει μόνο να χρηματοδοτούμε έργα που επιβάλλονται άνωθεν και δεν φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους ούτε καλύπτουν τους στόχους μας. Ο κύριος Πόλτσακ μίλησε επίσης για το σχεδιασμό. Βεβαίως συμφωνούμε και υποστηρίζουμε Ε, τους Δήμους και τις κοινότητες, γιατί πολύ συχνά οι μικροί Δήμοι ε, έχουν ανάγκες που δεν τις αναγνωρίζουν οι Βρυξέλλες. Ευχαριστώ την κυρία Μιχαήλοβα που μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω να ενώπιον σας να μιλήσω. Και σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητε μας, κύριε Φανίστε Ρόε, βεβαίως και θα προσκληθείτε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολλές από αυτές θα έχουμε και πυρογνώμονε που θα συμμετέχουν στι συζητήσει αυτές κτλ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ ε, τους ε, ερετούς εκπροσώπους του λαού. Εγώ ε, διατέλεσα επί μακρόν εθνικός βουλευτής και ξέρω ότι οι άνθρωποι που έχουν σαφή εντολή θα πρέπει να τα λένε έξω από τα δόντια να μιλάνε στα ράτα και οι ευρωβουλευτές έχουν τέτοια σαφή και ρητή εντολή από τους πολίτες τους τους ψηφοφόρους τους. Εγώ πάντα θα σέβομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ακούω τη γνώμη του. Η συζήτηση αυτή, καθώς επίσης και οι διμερείς συνομιλίες με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε τις προτεραιότητές μας, οι οποίες βασίζονται και στα όσα αποκομίσαμε από αυτές τις γόνιμες συζητήσεις με ευρωβουλευτές. Πέρα από το βασικό μας πρόγραμμα το οποίο σας έχει διανεμηθεί. Προσβλέπω λοιπόν αισιοδοξία στους επόμενους έξι μήνες. Θα είναι στενή η συνεργασία μας και ελπίζω γόνιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευγενικό τα λόγια σας για το Ευρωκοινοβούλιο, το εκτιμούμε και σας ευχαριστώ και για την ε, εισήγησή σας, για τις απαντήσεις που μας δώσατε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και αναμένουμε αυτή οι επόμενη έξι μήνες να είναι γεμάτη συνεργασία μεταξύ ημών. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διατάξη, όπου επόμενο σημείο είναι μια μελέτη που ζήτησε το θεματικό τμήμα Β σχετικά με τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διευθυντικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων μέσων της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 συνέργειες ανάμεσα στα διάφορα μέσα είναι απαραίτητες για να μην υπάρξει επικάλυψη και έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Συζητήσαμε αυτή τη μελέτη για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εθνικών και επενδυτικών ταμείων και των άλλων μέσων όπως το Horizon 2020, το EFSI ή το COSME already Είχαμε μια σχετική συζήτηση στο Κοινοβούλιο και θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε σήμερα τα πορίσματα για την τελική γνωμοδότηση που προετοιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών. Σήμερα ο κύριος Στέβαν Κά είναι εδώ μαζί μας και Με χαρά θα ακούσουμε την εισήγησή σας, ε, κύριε Κά. Thank you. Έχετε το λόγο. Thank you very much for the opportunity to... Uh, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη για τις συνέργειες που, που εκπονήσαμε στη διάρκεια των περισμένων έξι μηνών. Να πω δύο λόγια για το ποιοι είμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών είναι κομμάτι του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης Είμαστε κομμάτι ενός, ενός πολυεθνικού επιτελείου και λειτουργούμε εδώ και σχεδόν 40 χρόνια με εστιασμό στην πολιτική συνοχή, στην περιφερειακή πολιτική και όταν μιλάμε για συνέργειες είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η συνέργεια. Υπάρχουν και άλλοι όροι που είναι παρόμοιοι, αλλά που σημαίνουν όλα πράγματα. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε για συνοχή, ε, η συνέπεια που σημαίνει περισσότερο το να εξασφαλίζουμε την ε, συνοχή, τη λογική ανάμεσα στα προγράμματα. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε για συντονισμό, δηλαδή κοινέ πληροφορίε, κοινού πόρου κτλ. Αλλά ούτε και στην συμπληρωματικότητα, παραπληρωματικότητα που ένα είναι ένα ίσον δύο και μετά έρχεται το επόμενο επίπεδο. Έχουμε συνέργεια όπου ένα είναι ένα μα κάνει πάνω από δύο. Η συνέργεια αυτό σημαίνει. Και αυτό θα προσπαθήσω να σας δείξω με αυτές εδώ τις διαφάνειες για να δομήσουμε ότι όλες αυτές τις ε, πληροφορίες που συλλέξαμε σκεφτήκαμε ποιες τις προσπάθειες ε, που πρέπει να γίνουν για να δημιουργηθούν συνέργειες σε τέσσερις διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναρμονιστούν ε, οι ρυθμιστικές προδιαγραφές, μετά έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό που να είναι ευθυγραμμισμένος και τέλος χρειαζόμαστε εφαρμογή και σε σχέση με αυτό και την αναφορέ, αναφορές και το συντονισμό αυτών. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες δομές, διάφορα επίπεδα και διακυβέρνηση. Εδώ τώρα, μάλλον καλύτερα βλέπετε από τα φυλάδια που σας μοιράσαμε, εδώ βλέπετε περί τίνος πράγματος μιλάμε. Στην αρχή έχουμε κοινή διαχείριση. Έχουμε τα διάφορα ταμεία και μετά τα συγκρίνουμε με τα μέσα τα οποία, στα οποία υπάρχει άμεση διαχείριση. Έχουμε δομήσει το εμπειρικό τμήμα σε δύο στάδια. Πρώτα μιλήσαμε με διάφορους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επόμενο στάδιο συζητήσαμε με τους ανθρώπους στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τους όρους αναφοράς και το πρώτο, την πρώτη φάση διερεύνησης με την Κομισιόν και άλλους φορείς, επιλέξαμε έξι μέσα ή πλαίσια. Και από εκεί αναπτύξαμε έξι συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες όπου είδαμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη με βάση πού πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε παραδείγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τέσσερα μέσα, είτε πρόκειται για συσχετιζόμενα με τη χρηματοδότηση, μετά έχουμε δύο στατηγικά πλαίσια, ή δομές που προβλέπουν τον συνδυασμό, ε, δηλαδή τη συνέργεια ανάμεσα στις δύο πλευρές της εικόνας αυτής. Ε, προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε εδώ και την ανάπτυξη της υπαίθρου, την εταιρική σχέση για την ε, καινοτομία και εκεί και το Γεωργία ήταν ένα από τα στρατηγικά πλαίσια. Επίσης, θέλαμε να εξασφαλίσουμε την ε, κάλυψη, σχετικά καλή κάλυψη στις, για τις 28 χώρες. Δεν είχαμε πολύ χρόνο ούτε και χρήματα και γι' αυτό προσπαθήσαμε να εξετάσουμε όλα τα κρατημέλη, τα νέα κρατημέλη, ομοσπονδιακές δομές, πιο κεντροποιημένες δομές, μικρά, μεγάλα κρατημέλη και ελπίζουμε ότι έτσι με αυτές τις 7 περιπτωσιολογικές μελέτες καλύψαμε επαρκώς την Ένωση. Πρώτα όμως πρέπει να πάμε πίσω στο 2007 με 2013 το πλαίσιο 2007-2013 ε, περισσότερο χαρακτηριζόταν από τον διαχωρισμό και την ε, περιχαράκωση των μέσων ε, Ο εστιασμός δεν είχε δοθεί στις συνέργειες, αλλά είχε γίνει προσπάθεια να μην υπάρχει επικάλυψη, αλλά να υπάρχει και συμμόρφωση με τους κανόνες. Η επιδίωξη των ισορροπιών και θεματικά τονίστηκε το EDF ε, αλλά και όσον αφορά τις εδαφικά στα κάτι μέλη της περιφέρειας όπου υπάρχουν περιορισμένοι στόχοι συνοχής και ένας μικρός αριθμός εντοπισμένων ας πούμε στόχων τα πράγματα ήταν πιο εύκολο να επιτευχθούν. Επίσης για το 2007 με 2013 είδαμε τις βασικές προδιαγραφές, δηλαδή στρατηγική εφαρμογή, διακυβέρνηση και ούτω καθεξής. Τώρα, υπήρχαν διαφορετικά καθεστώτα, πράγμα το οποίο δημιουργούσε όμως περιπλοκό χαρακτήρα και αβεβαιότητα και γι' αυτό και οι φορείς εστιάστηκαν στην συμμόρφωση και όχι στη συνέργεια για τη διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση ήταν κατακαιρματισμένη στα διάφορα μέσα και στα διάφορα κονδύλια. Ωστόσο, προέκυψαν ήδη κάποιες πρωτοβουλίες για απαλή διακυβέρνηση. Ωστόσο, υπήρχε κατακαιρματισμός. Από την μια πλευρά είχαμε και για τα δύο μέσα, και για τις κοινή διαχείριση και τις ε, άμεσες διαχείρισης. κυρίως με την ατζέντα της Λισαβόνα και την Ευρώπη 2020 υπήρχαν γενικές στρατηγικές για συνέργειες, αλλά υπήρχαν κενά για συνέπειες, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ότι η, τα κονδύλια είναι πιο ε, στοχοθετημένα εδαφικά. Είναι σπάνιες λοιπόν οι συνέργειες επί τόπου. Ε, και επίσης ε, βλέπουμε ότι γίνανε προσπάθειες ε, δημιουργίας δυνατοτήτων, αλλά ανεπαρκώς. Δεν υπήρχαν συστηματικές προσεγγίσεις. Ας περάσουμε τώρα στο τρέχον πρόγραμμα 2014 με 2020. Οι, μετα... οι ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις είναι βασικές, αλλά παραμένουν κάποιες προκλήσεις. Οι κύριες ρυθμιστικές προόδοι που επιτρέπουν την επιδίωξη συνεργειών είναι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και ώστε με αυτό υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωση όρευση επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων σε κάποιο βαθμό. Υπάρχει δυνατότητα για ευθυγράμμιση των μοντέλων κόστους λόγω της αυξημένης χρήσης απλοποιημένων ε, μοντέλων και υπάρχει και ατζέντα απλοποίησης ε, όπου δημιουργήθηκε και το πρόσφατα το, ε, η ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση. Παρ' όλα αυτά, κάθε τομέα πολιτική εξακολουθεί να διέπεται από το δικό τη κανονισμό, πράγμα που δεν διευκολύνει τι συνέργειε. Ε, επίσης, η... δεν, δεν υπάρχει συνέργεια σε εθνικό επίπεδο και ε, το αριθμιστικό πλαίσιο είναι ήδη αρκετά περίπλοκο και οι συνέργειες το περιπλέκουν ακόμα περισσότερο. Έτσι μας είπαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε. Όλες αυτές οι αισθάσει είναι σημαντικές για την, για την κυβερνητική διακυβέρνηση μάλλον των προγραμμάτων, αλλά και για την εφαρμογή. Τώρα, στη διακυβέρνηση οι αλλαγέ είναι περιορισμένε και ε, ορίζονται από τι ρυθμιστικέ ανάγκε. Υπάρχουν πρωτοβουλίε σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει η ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση που την ανέφερα ήδη, διάφορε ε, οριζόντιες ομάδες εργασίας όπως η RTD, η ομάδα επαφή για τα δευτερικά ταμεία και διάφορε πρωτοβουλίε για τη στήριξη των κρατών μελών, για παράδειγμα Enterprise Europe και η πλατφόρμα Smart Specialization και σε επίπεδο 100 μελών γίνονται πρωτοβουλίες όπως ας πούμε το Ισπανικό Δίκτυο RTDR που στόχο έχουν να διερευνήσουν και να υλοποιήσουν συνέργειες όπου αυτό είναι δυνατόν. Το μοντέλο της κοινή διαχείρισης των ε, ταμείων είναι ήδη αρκετά περίπλοκο και αν προσθέσουμε και συνέργειες εκεί θα ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Τα νέα μέσα παραμένουν ε, μοιρασμένα ανάμεσα με θέματα και δραστηριότητες και σε επίπεδο της Κομισιόν, γιατί υπάρχει κατακαιρματισμός στο επίπεδο των γενικών διευθύνσεων, αλλά αυτό πρε... εστιάζουν στο προπαρασκευαστικό στάδιο και όχι στην εφαρμογή. Στα κάτι μέλη όμως, είναι αποκομμένες οι προσεγγίσεις, απομονωμένες η μία από την άλλη, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής. Σημαντική πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι μία πρόοδο για τη στατηγική ευθυγράμμιση. Κυρίω οι εταιρικέ σχέσει είναι ισχυρά δίκτυα για συνέργειε, τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πολιτική συνοχή, θεματική συγκέντρωση, ρεσιμότητα και επίση στρατηγικέ περιφερειακές είναι στοιχεία που βελτιώνουν την πολιτική συνοχή και συγκεντρώνουν διάφορους φορείς από διάφορες τομείς πολιτικής. Οι τομείς πολιτικής ε, μπορούν να επιτρέπουν ε, στην ε, Ε, συνέργεια ανάμεσα σε διάφορες ε, τομείς πολιτικής ε, και καλύπτουν πολιτικές και προτεραιότητες που εμπίπτουν σε διάφορα μέσα της Ένωσης. Τώρα, εταιρικές σχέσεις πρέπει να υπάρχει και εκεί ένα κεφάλαιο για το συντονισμό και για το πώς μπορούν να επιτευχθούν οι συνέργειες. Αλλά είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πρόκειται για συντονισμό και εδώ πρέπει να επανέλθουμε στην αρχή για τα διαφορετικά επίπεδα συνεργασία ή συντονισμού. Δεν αφορά συγκεκριμένα τη συνέργεια. Ε, και βεβαίω είναι περίπλοκο να υπάρξουν κοινέ στρατηγικέ για προγράμματα που μπορεί να ενσωματώνουν διάφορα κονδύλια, ταμεία και διάφορα μέσα. Τώρα, τι γίνεται στην εφαρμογή. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες ε, υπάρχουν κάποιε καλέ πρακτικές και μια από τις προκλήσει ήταν ότι ήμασταν πολύ νωρί στην προγραμματική περίοδο και είμαστε ήδη στο 2016 αλλά θα διαπιστώσετε θα μας έλεγε ο κόσμος ότι δεν μπορούμε να σα πούμε και πολλά γιατί δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε πολλά, είναι κάπως νωρί. Έχουμε λοιπόν δύο προοπτικέ. Η μία προοπτική είναι η, η, ε, τα, τα, τα, τα, ταμεία και τα διευθυντικά ταμεία και μετά έχουμε τα άλλα μέσα. Τι μπορούμε να κάνουμε από αυτή την προοπτική. Να κάνουμε ε, κοινέ προτάσεις, να κάνουμε κριτήρια συντονισμού ή κοινή συλλογή ε, στοιχείων και αξιολόγηση. Μπορούμε ενεργά να συνεργαστούμε με τις αρχές των επενδυτικών ταμείων, να διασυνδεθούν τα, τα οι δικτυακοί χώροι, να διοργανωθούν κοινά σεμινάρια ε, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αναφέρουμε και, να, είναι πράγματα που έχουν ήδη κάποιες φορές γίνει από πρωτοβουλίες. Η εικόνα όμως είναι άνηση. Εστιάσαμε στην προπαρασκευαστική βάση και όχι ακόμα στην εφαρμογή. Ωστόσο, είναι ένα ε, τομέα η προσεγγίση στα κατημέλη και ισχύουν πολύ διαφορετικές συνθήκες ε, ανάλογα με τον κάθε τομέα. Ε, από αυτό εξαρτάται η δυνατότητα εφαρμογής συνεργειών, ανάλογα δηλαδή με τις δυνατότητες και την εμπειρία των διαχειριστών κάθε φορά. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα σύντομα για τη διακυβέρνηση, τη στρατηγική εφαρμογή. Ε, στη Γερμανία υπάρχει ένα πολύ επίπεδο σύστημα εργασίας. Ξέρετε ότι έχουμε τα περιφερειακά ομοσπονδιακά κρατήρια και ομόσποδα κρατήρια συγγνώμη, και το ομοσπονδιακό επίπεδο. Και υπάρχει το θέμα της εφιούς ε, εξειδίκευσης. Συμμετέχει το ESI και το Horizon 2020. Στη Ρουμανία έχουμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για την πρωτοβουλία στη Γεωργία που έχουν ε, συσταθεί ομάδες εργασίας έτσι ώστε να εξεταστούν οι και οι συνέργειες ε, μέσα στο Ταμείο ε, το ΦΕΟΓΚΑ και στη Τσεχική Δημοκρατία ναι. υπάρχει μια δραστηριότητα, μια πρωτοβουλία ομαδική ε, που συμμετέχει το Ταμείο Συνοχής και το ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την έρευνα και την ανάπτυξη που έζησαν ε, το ορίζον 2020 και με αιτήσει από άλλες χώρες. Um, I Λίγες συστάσεις για να κλείσω και πάλι ακολουθώ τις τέσσερις διαστάσεις αυτές για τη ρύθμιση έχει σημασία να εναρμονίζεται και για τις κρατικές ενισχύσεις όπου είναι διαφορετικός ο βαθμός ε, της ανάγκης να συμμορφώνεται και επίσης ε, για τις αναφορές ακούμε ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται, τι συμβαίνει ε, στην άλλη πλευρά του λόφου. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για την κοινή χρηματοδότηση να έχουμε κοινέ προσπάθειες. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να συνδυαστούν οι πηγές χρηματοδότησης μόνο ορίζον 2020 και αυτό ε, μέχρι ενό βαθμού. Γιατί τη διακυβέρνηση επίσης έχει σημασία να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Μας το είπαν και οι ίδιοι. Δηλαδή δεν ε, παίρνουν ε, τις ίδιες προφορίες όλοι ανάλογα με το ποια γενική διεύθυνση θα ρωτήσουν. Και επίση είναι ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και με την ήπια διακυβέρνηση. Τώρα υπάρχει μια τάση να ε, ε, ε, επικεντρωνόμαστε στη συμμόρφωση. Δηλαδή να μην βάζουμε okay, σε διάφορα κουτάκια, αυτό δεν είναι διακυβέρνηση. Ε, στα στρατηγικά έγγραφα θα πρέπει να ξεπερνάμε το συντονισμό και τη συνεργασία, τι είναι η συνέργεια και πώς μπορεί αυτή να οριστεί και να επιτευχθεί. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε συμφωνίες εταιρικές, άλλες είναι πάρα πολύ λεπτομερείς και χαράσουν συγκεκριμένους δρόμους, άλλες είναι πολύ γενικόλογες, πέντε εκπροτάσεις και τελειώνει η υπόθεση. Θα πρέπει στην πράξη να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ομάδες εργασίας, ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά το πρακτικό στοιχείο λείπει μέχρι τώρα. Um, then finally implementation. Um, what would be good to see is joint work programs and joint calls. Κοινή προσπάθεια λοιπόν, κοινή συνέργεια, κοινέ επιτυχίες και επιτεύγματα, έτσι ώστε οι βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα να μπορούν να ε, εντοπίζονται κάθε φορά. Οι δικαιούχοι δεν γνωρίζουν κατά ανάγκη τα ωφέλη και τις ευκαιρίες που ανοίγονται με τις συνέργειες αυτές και είναι κρίμα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση γιατί τελικά η επιτυχία όλων αυτών των προσπαθειών θα εξαρτηθεί από τα όσα υλοποιούνται σε επίπεδο κρατών μελών επιτόπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διάφορες ε, επαφές και άτυπες και επίσημες. Πολλές φορές η συνεργασία γίνεται επειδή κάποιος γνώριζε κατά τύχη ναι, ναι, έναν άλλον άνθρωπο που είχε μια αντίστοιχη δραστηριότητα. Και πέρα από τις συνέργειες και τις συνδέσεις ε, θα πρέπει αυτές ε, να γίνουν πιο ελκυστικές. Γιατί μέχρι τώρα εμφανίζονται ως ένα πλέον βάσανο και πλέον, επιπλέον κόπος που δεν ήταν ο καθένας πρόθυμος να κάνει. Ή να υπάρχει ξεχωριστό κονδύλ του προϋπολογισμού ή ένα χρηματοδοτικό μέσο με μεγάλη μόχλευση για να γίνονται ελκυστικά όλα αυτά ή και η φήμη ξέρω εγώ, ένα σήμα αριστείας, μια σφραγίδα αριστείας, κάτι, μια βούλα. Και τέλος, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε όλα αυτά. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ελέγχει την πρόοδο. Ιδιαίτερα σε αυτό το πρώιμο στάδιο, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει στην πράξη για την περίοδο 2014-2020 και θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται επί τόπου, γιατί πολλές φορές μιλάμε για συνέργεια σε επίπεδο στρατηγικό και κεντρικό. και διάφορε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλό θα ήταν να ανταλλάσσουν απόψει, να έχουν και εκείνε μια τέτοια συνεργασία, ε, βέλτιστε πρακτικέ κτλ. Αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very, very Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τον συναδέλφος, Ο κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ. Από αυτά που άκουσα έτσι τα γρήγορα, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. πώς να το πω. Είναι κακός ο συντονισμός ε, ε, ανάμεσα στις Γενικές Διευθύνσεις Επιτροπής. Το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός. Αλλά καλό που το λέτε ξεκάθαρα. Και κάτι άλλο, από την προσωπική μου εμπειρία, Σουηδία. Η, συνέργεια ανάμεσα σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα είναι ε, μία πραγματικότητα που περιγράψατε. Τι γίνεται όμως ε, και με το συντονισμό χρηματοδοτικών μέσων με τα κράτη-μέλη, με τις περιοχές. Οι εθνικές αρχές μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ε, μια, ένα παρακαμπτήριο δρόμο σε μια τουριστική περιοχή και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Όμως, μπορεί να προκύψουν bottlenecks, συμφορήσεις. Και θέλουν κέντρα για να τα διαχειριστούν αυτό. και ζητάνε από τις περιοχές, από τα περιφερειακά ταμεία, από τα διαρθρωτικά ταμεία, να συγχρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα. Και άρα πρέπει να γίνει συντονιστός ανάμεσα στα εθνικά κονδύλια και τα τοπικά ευρωπαϊκά τελικά κονδύλια. Νομίζω και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας για την παρουσίαση. Εξαιρετική η παρουσίαση της μελέτης. Κρίμα που μας έρχεστε μόνο σήμερα να τα συζητήσουμε. Την περασμένη εβδομάδα το είχαμε στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Οπότε ε, και τα ψηφίσματα θα μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ εάν είχαμε ακούσει τη μελέτη προηγουμένως. Είναι εξαιρετική η μελέτη, επαναλαμβάνω, και ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε. Δύο σύντομες ειδικέ ερωτήσεις. Πρώτον, υπάρχουν μέσα όπως το multi-fund και το cross-funding έτσι, που βοηθούν κανονικά για τις συνέργειες, αλλά τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες δεν τα χρησιμοποιούν. Ζητώ συγγνώμη αν το είπατε και δεν το άκουσα και δεν πρόσεχα εκείνη την ώρα. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι μπορεί να βελτιωθεί εκεί ή τι κίνητρα μπορούν να δεθούν για να χρησιμοποιεί κανείς περισσότερο αυτά τα εργαλεία. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τη σελίδα 7 της παρουσίασής σας, σημείο 2, για το cross-cutting strategies, όπου αναφέρεστε στους στόχους του 2020 και θα με ενδιέφερε εάν τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και για τους πέντε στόχους του 2020 ή είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα ή παρατηρήσεις σας ανάλογα με το στόχο, ε, το κλίμα, την απασχόληση, την παιδεία και τους υπόλοιπους δύο. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις. Mm. Α, να θέσω εγώ δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, πολύ ικανοποιημένη δηλώνω από την έρευνα σας και την παρουσίασή σας, γιατί στην Ολομέλεια 1,5 λεπτό είχα να πω αυτά που ήθελα και προσπάθησα να πω ότι για τις συνέργειες θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλα τα διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα στα προγράμματα, και τα αποτελέσματά τους, αλλά και τους φορείς σε όλα τα επίπεδα. Οπότε ευχαριστώ που έχετε αυτή την πολυεπίπεδη προσέγγιση. Και δεν είναι ένα βήμα, πρέπει να βλέπουμε συνολικά τη διαδικασία. Με μία συζήτηση δεν εξαντλείται το θέμα ή ούτε και με μία μελέτη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε τα καλά παραδείγματα από διάφορα κράτη-μέλη. Επειδή τα κράτη-μέλη θέλουν να συνδέσουν τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα και τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, πιστεύετε πως ε, τα αποτελέσματα παρότι είναι περιορισμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή της θετικής πτυχής της ε, πολιτικής συνοχής και όλων των ε, εργαλείων. Προβολή της ιδέας της συνοχής, γιατί με τις συνέργειες αυτές είμαστε στον πυρήνα της πολιτικής συνοχής. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Um, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Για το πρώτο ερώτημα, για το συντονισμό ανάμεσα στις γενικές διευθύνσεις. Μπορεί να ακούγεται σκληρό. Αλλά μην δακτυλοδεικτούμε μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δακτυλοδεικτούμε γενικότερα. Είναι σημαντικό όμως να δούμε και τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Και το βλέπουμε στην έκθεση. Ένα θέμα είναι συντονισμό των γενικών διευθύνσεων, το άλλο είναι τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Και ο συντονισμό ε, ε, ο διατομεακό, ε, ούτω είπε. Μιλήσαμε με συναδέλφους από DigiGrow, Move, RTD, και υπάρχει προθυμία συνεργασία, Νομίζω θα βελτιωθεί η συνεργασία. Όλοι αναγνώρισαν ότι δεν είναι τόσο ε, ανικανοποιητική η μέχρι τούδε συνεργασία. Αλλά θα αλλάξει αυτό. Τώρα, ε, συντονισμός και ε, συνδυασμός ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ανεξαρτήτως πηγής και εθνικής χρηματοδότησης. Νομίζω ότι αυτό υπερβαίνει το αντικείμενο της μελέτης. Δεν μπορώ να επεκταθώ για αυτό το ζήτημα. Multifund και cross-financing programs. Ε, δηλαδή ε, πολλαπλά ταμεία, συνδυασμός ε, ταμείων και ε, διασταυρούμενη χρηματοδότηση. η αλληλεπίδραση της χρηματοδότηση από τα, τα ταμεία με, και συνδυασμό με άλλες μορφές χρηματοδότηση. Προσπάθησα να το εξηγήσω πέρσι, αλλά ήταν λίγο νωρί σε σχέση με την προγραμματική περίοδο. Δεν είχαμε δηλαδή πρακτικά παραδείγματα. Τον Ιούνιο παρουσιάσαμε τη μελέτη για τη στρατηγική συνοχή και τώρα έχουμε βρεθεί στο δεύτερο βήμα. Καλό θα ήταν για τις επιχειρήσεις πολλαπλών ταμείων να έχουμε επικαιροποίηση όσο περνάει ο καιρός. Για το 2020, πού να ξέρω, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ε, δείτε την FEE, αλληλέγγυη ανάπτυξη. Ναι, ε, όλα αυτά τα προγράμματα είναι ευφυής ανάπτυξη. Συνδυάζουμε αυτά τα ταμεία με τον ορίζοντα 2020. Είδαμε το κόσμο, είδαμε το ΕΦΣΥ, εξακολουθεί να είναι νέο, το ΣΕΦ. Και όταν τους ρωτήσαμε, όταν τους ρωτούσαμε ε, γιατί παντού εμφανίζεται το 2020, μας είπανε μα είναι ο μεγαλύτερος κορβανάς. Τώρα η δυσκολία αυτή σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα των ταμείων. Ορίστες 2020 και έτπα. Αυτά ήταν τα δύο βασικά και πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Ναι, εμέσως θα σας απαντήσω καταφατικά. Ναι, ευφυής ανάπτυξη. Τα καλά παραδείγματα μου είπατε από τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να τα βρούμε. Τα έχουμε βάλει ε, σε κατηγορίες στη μελέτη. Είναι πρόωρο, εφόσον μιλάμε για την εφαρμογή. Καλό παράδειγμα θα είναι να βρούμε μια ομάδα εργασία που τα συζητάει. Για θυμηθείτε ποια είναι τα τέσσερα επίπεδα τη ε, κανονιστική ρύθμιση, ε, ε διακυβέρνηση, στρατηγικό σχεδιασμό και, το, και Χρειαζόμαστε καλά προγράμματα και σε άλλες μελέτες υπάρχει τεκμηρίωση. Clean Sky. Όλοι αναφέρονται σε αυτό το παράδειγμα. Η πρωτοβουλία του ορίζοντα 2020 για τη δημιουργία δικτύου ε, για όσους έχουν λάβει με επιτυχία τη χρηματοδότηση. Άλλο ένα παράδειγμα από την Ουαλία. Ναι, ήταν αυτή που ήταν αρμόδια για το ΕΠΑ και για τον ΕΣΤΑ 2020. Δεν ασχολήθηκα εγώ με αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω. Αλλά είναι γείτονά μου, είναι στο διπλανό γραφείο. Οπότε ατύπω μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψει. Το θέμα είναι, γίνεται να μεταφέρουμε αυτές τις καλές πρακτικές από τον ένα τομέα στον άλλο. Σας ευχαριστούμε. Θα κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9. αύριο οι συντονιστές παρακαλούνται να παραμείνουν και θα συνεχίσουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Okay.